Παρακαλώ, θα ήθελα να καθίσετε όλοι για να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Äh, Πρώτος ε, τώρα ζήτησε τον λόγο ο κύριος Γκόλνης ε, επί προσωπικού. Κύριε Γκόλνης, πείτε μας παρακαλώ με βάση ποιο άρθρο του κανονισμού ζητάτε το λόγο επί προσωπικού. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για το άρθρο 164 επί προσωπικού διότι ενημερώθηκα ότι κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών ο Προεδρεύων, που ήσασταν εσείς κύριε Πρόεδρε, μετά από επίμονο αίτημα για διαδικαστικό, είπε ότι θα μπορούσε να μου δώσει ρεμιστικά αν δεν ησυχάσω. Ε, λοιπόν, Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό προς τα άτομό σας και προς ε, τη θέση σας, πρέπει να σας πω ότι αυτή η έκφραση μου φαίνεται πολύ περιφρονητική. Δεν ζητάω κυρώσεις κατά του βολευτή Σούλτς. Αναγνωρίζω ότι ο καθένας έχει ελευθερία έκφρασης εδώ. Όμως βάσει του άρθρου αυτού του κανονισμού θέλω να σας πω ότι το άρθρο 22 του κανονισμού για ε, τα καθήκοντα του Προεδρού, άρθρα 165 και 166 για τις πειθαρχικές αρμοδιότητες του Προεδρού, σας επιτρέπουν να διώξετε ή να επιβάλλετε κυρώσεις σε ένα βουλευτή ο οποίος ενοχλούσε σοβαρά την διεξαγωγή της συνεδρίασης, αλλά δεν είναι δυνατόν μετά, χωρίς να τον έχετε ακούσει καν, να διώχνετε έναν ευρωβουλευτή ο οποίος στη στιγμή που πήρατε την απόφαση αυτή δεν ενοχλούσε καθόλου τις συνεδρίες χωρίς προηγουμένως να τον έχετε ακούσει και χωρίς να του δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσει στις κατηγορίες που του προσάψατε. Νομίζω ότι όλα αυτά αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θέλει να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ που με ακούσατε, Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Γκόλνης. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της ε, Σουηδίας για την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρωθυπουργέ Λεφβεν, καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μας τιμή που σας ε, υποδεχόμαστε σήμερα για να μας πείτε τις απόψεις σας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν σας δώσω τον λόγο να υπενθυμίσω πως ε, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης δεν θα έχουμε διαδικασία και HDI ούτε μπλε κάρτες. Τον λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός της Σουηδίας. Παρακαλώ. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε Σούλτ, σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, κυρία Γεωργίευα, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, Ήταν η καλύτερη και η χειρότερη εποχή. Ήταν η εποχή της σοφίας, ήταν η εποχή της ανοησίας. Ήταν η εποχή της πίστης. Ήταν η εποχή του φωτός. Ήταν η εποχή του σκότους. Ήταν η άνοιξη της ελπίδας. Ήταν ο χειμώνας απελπισίας. Αυτά είναι τα αρχικά λόγια στο, στην ιστορία δύο πόλεων του Ντίκενς που περιγράφει την Ευρώπη στο τέλος του 18ου αιώνα. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να μιλάει και για τη σημερινή εποχή. Είμαστε πραγματικά σε... στο χειμών της απελπισίας. Οι εξτρεμιστές θέλουν να επιτεθούν στα θεμέλιά μας, η Ρωσία να μετακινήσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ένωσή μας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων, την κοινωνική απελπισία και την παγκόσμια προσφυγική κρίση. Όμως υπάρχουν και κάποιες ακτίδες ελπίδας. Η συμφωνία για το κλίμα, η παγκόσμια συμφωνία, οι νέοι βιώσι, ε, στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και οι τελευταίες, ε, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τις αφρικανικές χώρες που είναι πολύ καλύτερα. Αυτό δείχνει ότι η παγκόσμια συνεργασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και έχουμε και μια ελπίδα αν μείνουμε ενωμένοι απέναντι στην εξωτερική απειλή, αν αντιμετωπίσουμε μαζί τις κοινέ προκλήσεις με τη συλλογική μας δύναμη που απαιτείται για να τις επιλύσουμε. Εάν αντιμετωπίσουμε τα τελευταία εμπόδια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και χτίσουμε ξανά στεναρές κοινωνίες. Εγώ γεννήθηκα το 1957, την ίδια χρονιά με τη συνθήκη της Ρώμης. Η γενιά μου Είχε πολλαπλές ευκαιρίες και είχε πολλές ελπίδες για το μέλλον. Για πολλούς από εμά, ο κόσμος φαινόταν δικός μας για να τον εξερευνήσουμε, για να τον κάνουμε καλύτερο για το αύριο. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο καθήκον από το να δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες, την ίδια ελπίδα στους νέους της σημερινής εποχής. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι κινητήριος μοχλός για κάτι τέτοιο. Εάν ε, σταθούμε και υπερασπίσουμε την δημοκρατία, την ε, συνεργασία και την προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας. Αυτές τις βασικές ε, αρχές. Να ξεκινήσω με την δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή ενισχύουμε την κοινή μας δράση κατά της τρομοκρατίας τρομοκράτες που επιτίθενται με τον πιο δειλό και φρικόδη τρόπο κατά των κοινωνιών μας. Πολλές από αυτές τις ε, δράσεις είναι σκληρές, αλλά είναι απαραίτητε. Αλλά για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία πρέπει να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι ότι ορθώνουμε το, το ανάστημά μας, ότι υπερασπίζουμε τους Εβραίους πολίτες μας, τη στιγμή που αντισημιτικές απειλές, ε, μίσος και βία ακόμα μια φορά αντιχούν στην Ευρώπη μας. Είναι το να μην δεχτούμε ή το να μην διαδώσουμε ε, λαϊκίστικες, δημαγωγικές, εξτρεμιστικές, ακραίες απόψεις, ακόμη και αν ε, κερδίζουμε με φτηνό τρόπο το, τους πολίτες. Είναι το να υπερασπιστούμε τους ε, Ρωμά, ε, τους στοχούς. Η υπεράσπιση δημοκρατία σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε την ελευθεροτυπία, την δυνατότητα του να ενημερώνει κανείς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτική υποφελείται από το σωστό έλεγχο. Η υπερασπίση της δημοκρατίας σημαίνει είναι ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων σε μια για δίκαιη δίκη, το να μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην ε, κοινωνία, το να αγαπάνε όποιον θέλουν. Εάν δεν υπερασπιστούμε αυτές τις δημοκρατικές αξίες, θα χάσουμε την Ευρώπη, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και τώρα πάω στο δεύτερο σημείο, που είναι η συνεργασία. Πολύ σπάνια τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν μετακινηθεί στον πλανήτη όπως συνέβη σήμερα. Αλλά πολύ σπάνια και τόσο λίγες ευρωπαϊκές χώρες ε, βρέθηκαν έτοιμες να δράσουν. Πέρυσι το φθινόπωρο, τους δύο τελευταίους ε, δύο μήνες, η Σουηδία δέχτηκε 80.000 ανθρώπους. Αυτό ισοδυναμεί με 25 εκατομμύρια ετούντε άσυλο στην Ευρώπη συνολικά. Αυτό έφερε το σύστημα ασύλου μας στο χείλος του γκρεμού. Και εν απουσία ευρωπαϊκών λύσεων αναγκαστήκαμε να λάβουμε μονοσήμαντη μονομερή δράση. Η Συμφωνία Σέγγεν και η ελεύθερη κυκλοφορία που απορρέει είναι θεμελιώδης ακρογωνιαίος λήθος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικό στοιχείο της οικονομίας μας, για την οικονομία μας. Αλλά αν δεν αντιδράσουμε, μπορεί να χάσουμε αυτή την ελευθερία. Ακούω πολλά λόγια και σχέδια να προχωρήσουμε. Αλλά πολύ λίγη δράση, πολύ λίγα έργα. Και γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι και η ώρα να δράσουμε, να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου. Να εφαρμόσουμε την αναδιανομή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταπολεμήσουμε τη σωματεμπορία και να ενισχύσουμε την ε, κοινή εξωτερική πολιτική για να σταματήσουμε και να ανατρέψουμε τις αιτίε της ε, προσφυγικής κρίσης. Από το χάος πρέπει να περάσουμε στον απόλυτο έλεγχο, γιατί κινδυνεύουμε να υποσκάψουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία, υπό τη μορφή που την ξέρουμε τουλάχιστον. Με το βλέμμα προς τα εμπρός, προς το μέλλον, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν λειτουργεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν δεν δημιουργήσουμε μια νέα κοινή προσπάθεια, ένα κοινό σύστημα βιώσιμο για το άσυλο, όλο και περισσότερε χώρες θα δρουν μονομερό που θα ε, υποσκάψουν την κινητικότητα, το εμπόριο με αυτόν τον τρόπο και κυρίως τους ανθρώπους που φεύγουν, που μετακινούνται. Εμείς θέλουμε ω Σουηδία να υπάρξει ένα νέο σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δίκαιη κατανομή και όπου το άσυλο το ζητάει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τι μεμονωμένες χώρες. Πολύ πολύ απλά, εάν θέλουμε να μοιραστούμε τα εξωτερικά σύνορα και να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία στις χώρες μας, θα πρέπει να έχουμε το ίδιο σύστημα υποδοχής, το ίδιο σύστημα ασύλου. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο κοινό σύστημα ασύλου μπορούν να συμμετέχουν στην συνεργασία Σέγγεν. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Και τώρα πάω στο τρίτο σημείο. Την προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας. Δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά για να παραμείνουμε ενωμένοι ε, για να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα παράπονα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντού, σε όλη την Ήπειρο, δεν θα πρέπει να τα παραβλέψουμε. Αυτά τα παράπονα δείχνουν την τρομακτική ανάγκη να τονίσουμε τι είναι αυτό που μας κρατάει μαζί. Το ευρωπαϊκό πνεύμα, ε, τη συνεργασία, ε, την ευρωπαϊκή για τους πολίτες. Θα πρέπει να δείξουμε την αξία που έχουν 28 ε, χώρες και οι 500 εκατομμύρια πολίτες από κοινού για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή που σε καμία χώρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει σε αυτή την περίπτωση παγκόσμιας αλληλεπίδρασης, να δημιουργήσουμε ακόμα μια, μεγαλή, μια ακόμα ε, πιο μεγάλη αγορά και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας ε, αναστάτωσης. Αν όμως η ευρωπαϊκή συνεργασία θα αποκτήσει αυτή την ευρεία, την πλατιά υποστήριξη που χρειάζεται στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να έχουμε μια ένωση η οποία κάνει πολύ περισσότερα για την ευημερία των λαών της, των πολιτών της. Σε έναν κόσμο όπου 62 άτομα έχουν στο έλεος τους 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους όταν 62 άνθρωποι έχουν όσα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε πλούτο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, να υπάρχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη του κοινού. Γιατί όταν ο κόσμος και οι επιχειρήσεις ενισχυθούν, αναπτύσσονται οι οικονομίες. Σε μια κοινωνική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός υπερασπιστής των καλών ε, εργατικών συνθήκων για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι εργαζόμενοι δεν αναγκάζονται ε, να ανταγωνιστούν ε, ο ένας τον άλλο για... σε μια κούρσα προς τα κάτω γιατί πάντα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια στον τόπο εργασίας. Θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιοποιηθεί το δυναμικό της ε, εργατικής, του εργατικού της δυναμικού. Εάν κάνουμε αυτές τις προσπάθειες μπορούμε να αυξήσουμε μέχρι το 2030 το ΑΕΠ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 12%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δράσει μόνο ως κέντρο για υγιή δημοσιονομικά, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και για μια ισότιμη θέση όλων στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι και ηθικά σωστό και οικονομικά έξυπνο. Σε μια κοινωνική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει συλλογική δράση κατά της ανεργίας των νέων που υποσκάπτει και την νεολαία της και τις οικονομίες αλλά και την πίστη της κοινωνίας μας για το μέλλον. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε επενδύσεις για την εκπαίδευση, να επεκτείνουμε τις ανταλλαγές των Ευρωπαίων φοιτητών όχι με, μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην, στο Λύκειο και να δημιουργήσουμε τις θέσεις απασχόλησης για το μέλλον, για τους νέους. Ε, είναι κοινωνική επένδυση αυτή να έχουμε φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες και μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτή είναι η κοινωνική Ευρώπη, η οποία μπορεί να κερδίσει τον κόσμο στην Ευρώπη. Η πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση της οδηγίας για την ε, απόσπαση των εργαζομένων ε, δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια ε, για να κινηθούμε προς τα εκεί το να έχουμε πιο αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο. Αυτά είναι εκ των όνου κάνευ. Α συνεχίσουμε λοιπόν προ τα εμπρό, προ τα πάνω. Α κάνουμε μια προσπάθεια προ την κορυφή και α φτιάξουμε μια στρατηγική για να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική Ευρώπη. Και αν γίνει μια τέτοια σύνοδο κορυφή που θα γίνει το 2017, εγώ με μεγάλη χαρά και τιμή θα την διοργανώσω. Βουλεύουμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξυπηρετεί και τις αγορές, ναι, αλλά ακόμα περισσότερο την ευημερία των πολιτών της. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν είναι βασικοί φορείς ε, για να προωθήσουν αυτά τα τρία βασικά θέματα που σας ανέφερα. Για να καλύψουμε αυτό το κενό στην Ένωσή μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ίδια ελπίδα που εγώ έζησα, εγώ και η γενιά μου, η γενιά του 1957 και η γενιά του 1997 και του 2007 και του 2017 και οι επόμενες ακόμα γενιές για να μπορέσουν να ζήσουν την ε, ίδια ελπίδα. Ούτως ώστε αυτή, αυτός ο χειμώνας της απελπισίας της Ευρώπης, ο οποίος ήταν μακρύς, να σταματήσει. Αν όμως ε, υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τις πιο δύσκολες στιγμές της, Εάν τα λόγια τα κάνουμε πράξη για να αντιμετωπίσουμε την ε, μεταναστευτική κρίση, αν δημιουργήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη που αυξάνει την ευημερία των πολιτών καθημερινά, στην καθημερινότητά τους, τότε μόνο θα είμαστε σε θέση και στις καλύτερες εποχές και στις χειρότερες εποχές να δημιουργήσουμε μια νέα άνοιξη ελπίδα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Γεωργίευα, την πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω σε αυτήν την συζήτηση και να σας ε, διαβιβάσω τους χαιρετισμούς του. Πράγματι είναι η χειρότερη και η καλύτερη καιρή, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο καιρός και η στιγμή στην Ευρώπη να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να υψώσουμε το ανάστημά μας. Και χαίρομαι που σας καλωσορίζω κύριε Πρωθυπουργέ στην αίθουσα αυτή, εδώ όπου αυτό ακριβώς μόλις κάνατε. Σας ευχαριστώ. Η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία διαμόρφωσε τη μοίρα της με αξίες και την πεποίθηση ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μια δίκαιη κοινωνία. Και έχετε επηρεάσει και χώρες ε, πέρα από τα σύνορά σας, ε, την υπόλοιπη Ευρώπη. Να υπενθυμίσω πως ε, με τους σκανδιναβούς εταίρους σας, εσείς ήσασταν οι πρώτοι που αντιληφθήκατε την αξία της ελεύθερης μετακίνησης, γιατί το Σκανδιναβικό Συμβούλιο του 1950 ήδη ξεκίνησε με μια περιφερειακή αγορά εργασίας ε, και είναι κάτι το οποίο βεβαίως βοήθησε και εσάς και την Ευρώπη. Σήμερα, εξ ονόματος ε, του Προέδρου μας, ε, θα ήθελα να επενέσω την Σουηδία για την αντίδρασή της στη μεταναστευτική κρίση. Η χώρα σας εδώ και καιρό λαμβάνει αναλογικά τον υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που αναζητούν προστασία. Πολύ πριν ξεκινήσει η τωρινή κρίση και πραγματικά είστε φάρος φωτεινός. Όταν μια χώρα τόσο βόρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται τόσο άμεσα από τα γεγονότα στον Νότο, γνωρίζουμε ότι είναι κοινή η μοίρα. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της και καμία χώρα δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Σουηδία, ούτε η Αυστρία, ούτε η Γερμανία. Καμία χώρα δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μόνη της. Μαζί πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Μαζί πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εξαρτώνται από μας για την επιβίωσή τους. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχει κάνει η Σουηδία και αναστήλαμε τη μετεγκατάσταση προσφύγων στη Σουηδία από Ελλάδα και Ιταλία. Είναι ρεαλιστικό και δίκαιο σήμερα όπως είπατε, πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη στην Ευρώπη, να αποκατασταθεί το σύστημα Σέγγεν. Η χώρα σας γνωρίζει το τι σημαίνει το να μην υπάρχει Σέγγεν και εντυπωσιάστηκα από το πόσο κοστίζουν η έλεγχη στη γέφυρα Όρεσουντ που συνδέει τη χώρα σας με την Δανία. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα. Την Παρασκευή που μας πέρασε η Κομισιόν δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη για τα βήματα αποκατάστασης της ε, Σέγγεν και για να έρθουν όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι μέχρι το τέλος του έτους το αργότερο. Έτσι έχουμε την δυνατότητα να γίνει πιο ανθεκτική η Σέγγεν και πρέπει να διδαχτούμε από την κρίση αυτή, πως το σύστημα λειτουργεί μόνο εάν συμμετέχουμε όλοι. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Και προφανώς πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε. Στην Κομισιόν δεν μας ενδιαφέρει τώρα να κατηγορούμε, μας ενδιαφέρουν οι λύσεις, να στηρίξουμε όλα τα κράτη-μέλη για να σηκώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί για να αποκαταστήσουμε και να προστατεύσουμε την Σέγγεν. Να αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρωθυπουργέ, που αναφέρατε Επίσης ένα θέμα αξιών στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι ένα μεγάλο επίτευγμα πολύ περισσότερο από έναν τρόπο οργάνωσης της οικονομίας είναι το τι είμαστε, είναι κομμάτι των συνθήκων μας και της ταυτότητάς μας. Η Σουηδία έχει γράψει κεφάλαια ολόκληρα της ιστορίας αυτής. Ε, ακούγοντάς σας, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ε, βλέπω πως εξακολουθείτε να γράφετε κεφάλαια σε αυτή την ιστορία. Δείξαμε λοιπόν στον υπόλοιπο κόσμο πως η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να έχει ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη χέρι-χέρι. Ο πρώην εργοδότης μου το 1900, ε, το, ο πρώην εργοδότης μου Παγκόσμια Τράπεζα είχε αποκαλεί στην Σουηδία μια υπερδύναμη του τρόπου ζωής ε, και πραγματικά εσείς είστε αυτοί οι οποίοι δημιουργείτε τα πρότυπα όσον αφορά τη σχέση των δύο φίλων, την ισότητα και το κράτος πρόνοιας. Και ακριβώς ε, η πρόκληση τώρα είναι να προσαρμοστούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όταν εμείς γεννηθήκαμε. Έχοντας αυτά κατά νου, η αναγκαιότητα συνεχούς ε, προσαρμογής είναι αυτό που μας οδήγησε στην Κομισιόν να ξεκινήσουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ορίζει αρχές και πρακτικές για να διασφαλίσουμε πως ε, η δουλειά θα είναι αξιοπρεπής και δίκαια, θα έχουμε ίσες ευκαιρίες, δίκαιες συνθήκες και επαρκή κοινωνική προστασία. Για να υπάρχει δικαιοσύνη για τα άτομα, αλλά να υπάρχει και μια ελαστικότητα και ευελιξία στην αγορά εργασίας και στην οικονομία μας. Αποκαλύπτοντας λοιπόν τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία θα αποκαλυφθούν τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Να τελειώσω λέγοντας τα εξή. Εδώ και πολλές δεκαετίες η Σουηδία ενσάρκωνε τις ευρωπαϊκές αξίες. Τις αξίες της ισότητας, της ανθρωπιάς, για τους ανθρώπους που αναζητούν προστασία. Και σήμερα αποδείξατε πως είναι πολύ ισχυρές αυτές οι αξίες. Θα απαντήσουμε λοιπόν στη μεγαλύτερη αυτή πρόκληση της γενιάς μας. Οι αξίες αυτές είναι το φως που πρέπει να ακολουθούμε. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή λύση και είναι η μόνη λύση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπουργέ και να ευχαριστήσω και την Σουηδία που είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της λύσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριο Χέκμαρκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Είναι καλό να ακούμε τον Πρωθυπουργό μας να μιλά έτσι ξεκάθαρα εκ μέρους της Σουηδίας και να λέει ότι η Σουηδία πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ζούμε σε καιρούς όπου οι κρίσεις μας έρχονται απ' έξω. Έχουμε διάφορες κρίσεις. Το Ντάες, Συρία, τρομοκρατία, έχουμε την κλιματική αλλαγή διάφορες κρίσεις και εκείνη των προσφύγων βέβαια και των ετούν τον άσυλο. Φυσικά λοιπόν είμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις. Μόνο μέσα από μια ισχυρή Ευρώπη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε ότι μπορούμε όλα αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουμε την επόμενη εβδομάδα για παράδειγμα μόνοι μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε, να επικεντρωθούμε στην συνεργασία. Τη χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Και αυτό γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά και διαφορετικά προβλήματα και σίγουρα η λύση είναι πολύ καλύτερη αν έρχεται από πολλούς μαζί από ότι από έναν. Η Ευρωπαϊκή... Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας, αλλά πιο πολύ να αναρωτιόμαστε τι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι τώρα και στο κοινωνικό. Δεν πρέπει να αποδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία παίζοντας αυτό το παιχνιδάκι ζητημάτων που περνάνε από τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Τούμπαλιν. Οι πολίτες στην Ευρώπη διαμαρτύρονται και το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και εμείς αυτό στην Σουηδία ότι έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία. Πρέπει να μειωθεί. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ. Να επικεντρωθούμε στην μείωση της γραφειοκρατίας για να μπορούμε να δρούμε καλύτερα, ε, να κοιτάξουμε και τη σταθερότητα των οικονομιών μας και να φροντίσουμε να μιλάμε εκ μέρους του κομματό μας γιατί μερικές φορές λέμε ότι θέλουμε να ξοδέψουμε χρήματα αλλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Οι πρόσφυγες φυσικά είναι μια τεράστια κρίση κατανομή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, τηρώντας τους κανόνες. Και στην γέφυρα εκεί όπου επανήλθαν οι έλεγχοι, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, και να δούμε τι γίνεται γενικότερα με τις μεταφορές. Αν υπάρχουν οι πρόσφυγες, όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όλες οι χώρες. Ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ε, ευθύνες της. Για την ε, Τουρκία υπήρχαν κάποιες απαιτήσει για την ελευθερία του τύπου, για παράδειγμα. Σε αυτά πρέπει να επιμείνουμε. Θέλουμε μια Τουρκία περισσότερο δημοκρατική, που να ανταποκρίνεται περισσότερο στο κράτος δικαίου. Εδώ πρόκειται για τις ζωές ανθρώπων, ανδρών και γυναικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ισχυρή και για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλές προσπάθειες για πολύ καιρό και τις προσπάθειες αυτές θα τις κάνουμε μαζί από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτέλα για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, η όλο πάθος ομιλία σας με εντυπωσίασε. Μιλήσατε για δημοκρατία και συνεργασία. Μιλήσατε για αξίες. Για να κερδίσουμε τη μάχη για το μέλλον της Ευρώπης δεν πρέπει να παίξουμε στο στρατιωτικό πεδίο. Ούτε στη Συρία ούτε αλλού. Η μάχη για την Ευρώπη είναι μάχη αξιών πάνω απ' όλα. Θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιους μετασχηματισμούς των τελευταίων δεκαετιών χωρίς να υποσκάψουμε αντίθετα ενισχύοντας τις αξίες μας. Και υπάρχει ιδίω μια αξία που είναι πιο σημαντική από όλες. Αυτή της αλληλεγγύης. Σήμερα η Ευρώπη πλήττεται από εγωισμούς και εθνικισμούς. Ίσως πια λοιπόν δεν είναι της αυτή η λέξη και όμως είναι θεμέλιο της Ευρώπης. Αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Ο Ούλοφ Πάλμ ε, πίστευε σε αυτές. Και πριν από λίγες μέρες ε, πέρασαν, γιορτάσαμε τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Να σας θυμίσω μία φράση του. Έλεγε ο Πάλμ. Για μας η δημοκρατία είναι ένα θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι η πολιτική ελευθερία. Αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη σημαίνει καταρχάς αλληλεγγύη απέναντι στον κατατρεγμένο που φεύγει από τους πολέμους. Μιλήσατε για 80.000 ε, πρόσφυγες που δεχτήκατε εσείς στην Σουηδία. Ευχαριστούμε, Πρωθυπουργέ. Και πιστεύω ότι Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση τα κράτη από μόνα τους δεν μπορούν να τα καταφέρνουν. Η Γερμανία από μόνη της δεν μπορεί, η Σουηδία από μόνη της δεν μπορεί. Χρειάζεται ένα κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου το οποίο θα συνοδευτεί από μία αναθεώρηση του Δουβλίνου, όπως είπατε και εσείς. Αλληλεγγύη σημαίνει να υπρασπιστούμε την κοινωνική Ευρώπη, που πολύ σωστά υπενθυμίσατε, ότι δεν κάνει διαιρέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους, αλλά που τους ενώνει και τους προστατεύει όλους. Αυτό σημαίνει αναγνωρίζει σε όλους τους εργαζόμενους, όποια και είναι η εθνικότητά τους, ε, τον ίδιο μισθό για την ίδια εργασία. Στην ε, ομάδα μου και χάρη στη σημαντική συνεισφορά της ε, αντιπροσωπείας της χώρας σας, πετύχαμε να διατηρήσουμε τη δέσμευση της Επιτροπής ε, Juncker απέναντι στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Το χαιρετίζουμε αυτό και δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η προσπάθεια με όλες τις σημαντικές ε, εξελίξεις που έπονται και που απορρέουν ουσιαστικά από αυτή τη σημαντικότατη οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ECR, ο κύριος Χένκελ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πριν από τρεις εβδομάδες μιλούσαμε στο Στρασβούργο για δύο βουλευτές οι οποίοι μίλησαν εκτός της αιθούσης για διαταγές ε, που εδόθηκαν για να ανοίξουν άνθρωποι πυρ θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ε, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τις 19 ε, Μαρτίου θα έχουν εγκαταλείψει την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Κύριε, κύριε Πρωθυπουργέ, ε, είπατε δύο φορές πως γεννηθήκατε το 1957. Εγώ τότε πήγα με το ποδήλατο στο Γκέτεμποργκ και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η χώρα σας. Κοιτάξτε, ε, θα σας πω για ποιο λόγο είναι ευτυχής η χώρα σας. Πρώτα απ' όλα δεν μπήκε στο ευρώ. Το 1989 ως πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Βιομηχάνου με είχαν καλέσει στο εμπορικό επιμελητήριο τη Στοκχόλμη για να μιλήσω για το ευρώ, αλλά ευτυχώ ο Σουηδικό λαό ήταν εξυνότερος και από εμένα και από τους Σουηδού ε, βιομήχανου. Και εμεί στη Γερμανία αν ψηφίζουμε για κάτι είναι για το εάν θα χτίσουμε κάπου ένα σειροδρομικό σταθμό. Και βλέπουμε λοιπόν πως σε διάφορους δείκτες, είτε μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, είτε για ανεργία, η Σουηδία πάει καλύτερα από την Ευρωζώνη. Εσείς λοιπόν δείχνετε όχι μόνο στους αλλημοκράτες φίλους σας, αλλά σε όλους τους ευρωρομαντικούς, πως ε, ένα νόμισμα δεν ε, μπορεί να ε, υποκαταστήσει την δημοσιονομική κουλτούρα της κάθε χώρας και πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτήν και δεν μπορεί όλες αυτές οι διαφορετικές δημοσιονομικές κουλτούρες να υπαχθούν σε ένα νόμισμα. Δείχνεται πως το μικρό μπορεί να είναι όμορφο και δείχνεται επίσης πως η Ευρώπη δεν υποφέρει από την έλλειψη περισσότερης Ευρώπης αλλά από την υπερβολική Ευρώπη. Επίσης, δεύτερον, είστε ευτυχείς στην Σουηδία γιατί έχετε μια υπεύθυνη πολιτική ε, για το άσυλο. Ως μέλος της ε, Διεθνούς Αμνηστίας ξέρω πόσες δυσκολίες έχετε τώρα για να ελέγξετε τα σύνορά σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, η κατάσταση δεν είναι ανευθυνότητα αυτό το οποίο σας χαρακτηρίζει, ήταν υπευθυνότητα αυτό το οποίο κάνατε. Από τους ε, ετούντες άσυλο των τελευταίων ετών 72,3% ήταν άντρες και βλέπουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα σε διάφορες πόλεις όπως την Κολονία. Όμως έχει σκεφτεί κανείς από σας τι σημαίνει όταν αυτοί οι άντρες θα φέρουν εδώ πέρα τις ε, γυναίκες τους ή το τι σημαίνει ότι άφησαν εκεί πέρα μόνες ανυπεράσπιστες τις γυναίκες και τις αδερφές τους. Οι άνθρωποι επίσης αυτοί δεν έρχονται μόνο από εμπόλεμες περιοχές, αλλά από άλλες περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ ασφαλείς. Έχει σκεφτεί κανείς πόσοι άνθρωποι κινδύνευσαν ή έχασαν τις ζωές τους γιατί ακολούθησαν την πρόσκληση που τους απίφθινε η γερμανική κυβέρνηση και πίστεψαν ανεύθυνους διακινητές. Και έρχομαι εδώ πέρα στον τρίτο λόγο για τον οποίο είναι ευτυχής η Σουηδία στο ευρώ και στην ε, πολιτική την προσφυγική η γερμανική κυβέρνηση δεν έφερε σε αδιέξοδο μόνο το γερμανικό λαό αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αντίθεση με αυτό η Σουηδική κυβέρνηση ασκεί υπεύθυνη πολιτική. Το ότι τώρα η χώρα σας ε, έχασε την ε, θέση της ηθικής υπερδύναμης από τη Γερμανία της Μέρκελ δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Αντιθέτως θα πρέπει οι Γερμανοί μάλλον να μην είναι τόσο περήφανοι για αυτή την αμφίβολη τιμή. Σα ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους τον λόγο έχει η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Πρωθυπουργό. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι θετικό που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Η Σουηδία το γνωρίζουμε καλά όλοι. Είναι μια χώρα μέλους μεσαία όσον αφορά το μέγεθός της, τη δύναμη της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρωθυπουργέ όμως, προσοχή, αυτή τη δυνατότητα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Αναφερθήκατε στη Συμβασία του Δουβλίνου, Είπατε ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική ασύλου που να λειτουργεί καλά και γι' αυτό χρειάζεται να την μεταρρυθμίσουμε. Να συνεργαστείτε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε καλύτερη ακόμα συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Επίση, κύριε Λεύνεν, θέλω να σα ρωτήσω και το εξή. Τι γίνεται με το Συμβούλιο τη Ευρώπη, προσπαθήστε, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Προσπαθήστε να πείσετε τους συναδέρφους σας για να έχουμε μια πραγματική μεταναστευτική πολιτική και για να προχωρήσουμε στην αλλαγή αυτή που χρειαζόμαστε. Είδαμε τι έγινε μέχρι τώρα. Η Σουηδία έχει αλλάξει πολύ. Τώρα προσπαθεί να κερδίσει σε αξιοπιστία. Πρέπει να πείσουμε και άλλες χώρες να προχωρήσουν. Επίσης, η χώρα μας είναι μια χώρα που θεωρείται αρκετά παθητική απέναντι σε όλες αυτές τις ροές. Ναι, αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Μόνο έτσι, μόνο αν όλοι αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εντάξει, για την ε, Τουρκία αυτό που αποφασίσαμε δεν θα λύσει το πρόβλημα τελικά γιατί πάρα πολλά πράγματα βρίσκονται σε κρεμότητα και πάρα πολλά αντιβαίνουν σε συνθήκες, στην Σύμβαση της Γενέβης κλπ. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν έτσι καλώς να έρθουν στην Ευρώπη, θα το κάνουν όπως και να έχει το πράγμα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την κοινή πολιτική μέσω της οποίας θα αναλάμβαμε όλοι τις ευθύνες μας. Αν υπήρχε δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε να επαναληφθεί η ελληνική τραγωδία και να μην ξαναδούμε τα ίδια σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το θέμα λοιπόν το προσφυγικό δεν θα λυθεί μέσω της Τουρκίας. Βρείτε άλλες λύσεις, βρείτε νόμιμους τρόπους για να φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Ας έχουμε ένα σύστημα ασύλου υπεύθυνο που θα επιτρέπει και την κατανομή των προσφύγων δίκαια μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών. Η λύση με την Τουρκία δεν θα λειτουργήσει. Χρειάζεται μια κοινή πολιτική ασύλου. Αναλάβετε τώρα μια τέτοια πρωτοβουλία κύριε Πρωθυπουργέ και πείστε και τους συναδέρφους σας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε. Δείξτε ότι είσαστε πραγματικά ηγέτης, ότι έχετε τέτοιες ικανότητες ηγετικές. Δείξτε εσείς το δρόμο. Πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί θέλουμε διαφάνεια στις εργασίες μας. Το ίδιο να ισχύσει και στο Συμβούλιο. Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης δεν πρέπει να είναι αντίθετος αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε για να λειτουργήσουμε επικοδομητικά. Η Ευρώπη αξίζει πολύ περισσότερα από όσα έχουμε μπορέσει να κάνουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Για την Ενωμένη Αριστερά, η κυρία Μπιόρκ. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Σουηδία ανέλαβε τις ευθύνες της το 2015 και υποδέχτηκε μία σειρά από άτομα τα οποία έφευγαν από τόπους πολέμου. Είδαμε τι συνέβη το φθινόπωρο, είδαμε την απόφαση να κλείσουμε τα σύνορά μας. Ήταν η καλύτερη δυνατή απόφαση, δεν το ξέρω, δεν το συζητήσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίσουμε τις ίδιες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό τώρα πια επίπεδο. Θα πρέπει να υποδεχτούμε αυτά τα άτομα με οργανωμένο τρόπο ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κλείσουμε τα σύνορά μας ούτω ώστε να έχουμε τον χρόνο να πνεύσουμε λίγο. Τι θα συμβεί. Για μένα ήταν και είναι ξεκάθαρο, ε, Πρωθυπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποδεχτεί μια σειρά από ανθρώπους Μπορούμε να μιλήσουμε για το αν είναι μεγάλο το νούμερο, μικρό το νούμερο, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να παίξει η Σουηδία ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει τα σύνορά τη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν βλέπουμε τη σωστή στάση στο Συμβούλιο. Έχουμε θέμα ε, του τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη με μια αστυνομία δική της ε, που θα δράσει σε, τρίτη, σε τρίτες χώρες ε, που θα έχει περιπολίες στη Μεσόγειο και αυτή δεν είναι λύση. Ούτε η συμφωνία με την Τουρκία είναι λύση. Οι πρόσφυγες δεν είναι ψάρια, δεν είναι ποσοστώσεις, είναι άτομα. Άτομα τα οποία έχουν ψυχή, έχουν καρδιά, έχουν συναισθήματα, έχουν σάρκα και οστά. Δεν είναι αντικείμενα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε μαζί να δράσουμε συντονισμένα. Είδαμε ότι έκαναν οι μεν και οι δε στην Ευρώπη. Πρέπει να πάρουμε και ηθική στάση, αλλά θα πρέπει να έχουμε και πολιτική στάση. Θα πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο εναλλακτικό, θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε ρεαλιστικά. Τι τελευταίες μέρες έγιναν συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ λίγες. Έπρεπε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Τώρα, τι πρέπει να, κάνουμε όσοι τι πρέπει να κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες, τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, τι πρέπει να... και τι μπορούμε να προσφέρουμε στους πρόσφυγες. Θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας, αλλά και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι στο Συμβούλιο. Πρέπει να δούμε τώρα, το 2016 τι θα είναι. Θα είναι η χρονιά αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες ή θα είναι μια χρονιά που θα υψωθούν και άλλοι τύχοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς, την πρόεδρος των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το ότι φέρατε έναν ήρεμο τόνο στην συζήτηση και στην αντιπαράθεση αυτή για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Αν σκεφτούμε τη συζήτηση την σημερινή, την πρωινή εννοώ, νομίζω πως λίγη περίσκεψη θα μας ωφελήσει όλους, αν σκεφτούμε το τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Επίσης να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τη Σουηδία, τη χώρα σας, γιατί κατά την άποψή μου, εσείς εδώ και καιρό έχετε την καλύτερη πολιτική για τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο στην τωρινή κορύφωση του τελευταίου έτους, και όταν επαναφέρατε τους συνοριακούς ελέγχους, τότε η εντύπωσή μου ήταν πως τώρα να το χτυπάει το καμπανάκι από τη Σουηδία. Η Σουηδία λέει δεν μπορούμε άλλο, πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά θέλουμε παρόλα αυτά μια ευρωπαϊκή λύση. Ε, βεβαίως η αναζήτηση αυτής της ευρωπαϊκής λύσης ε, εξακολουθεί να αργεί. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε ακόμα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Έχουμε παγκόσμιες αλλαγές και παγκόσμιες προκλήσεις. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κανεί την εντύπωση ότι ο χρόνος είναι άπειρος. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε πως μια ομάδα κρατών θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά στην πολιτική των προσφύγων και να πει πως εμείς είμαστε αυτά τα κράτη που είναι διατεθειμένα μεταξύ μας να φροντίσουμε αλληλέγγυα για την υποδοχή περισσότερων προσφύγων. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε με την Τουρκία εντάξει, είναι αντικείμενο αλλά πού θα βρεθούμε εάν βρεθούμε στην διαχείριση του εξωτερικού συνόρου Ελλάδας-Τουρκίας και το μόνο που κάνουμε είναι να μοιράζουμε ανθρώπους. Λοιπόν, είπατε επίσης πως θα πρέπει να μυθούμε απέναντι σε νέους φόβους ε, όταν ε, δεν ζητάτε εσείς συγγνώμη για την εισαγωγή του ευρώ, δεν ξέρω, του ευρώ δεν ξέρω τι πρέπει να πει εδώ πέρα ο πρώην πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων. Αλλά μία πραγματική αμαρτία που υπάρχει εδώ πέρα για την οποία πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη είναι η ίδρυση του κόμματός σας της εναλλακτική για τη Γερμανία γιατί έτσι επιδεινώθηκε το κλίμα του φόβου. Οι Ευρωπαίοι, κυρίες μου και κύριοι, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αρχίσουν να φοβούνται όταν δεν είναι πλέον σε θέση να δρουν από κοινού απέναντι σε παγκόσμιες προκλήσεις ε, που όθησαν τους πρόσφυγες προς τα εμάς και εμείς προσπαθούμε να τους αποθήσουμε. Για αυτή την κοινή δράση πρέπει να μιλήσουμε. Η απέτηση προς τις ε, πλουσιότερες και σταθερότερες χώρες του κόσμου θα είναι όλο και πιο έντονη. Χτες ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τους ε, πρόσφυγες μας είπε ποια είναι η παγκόσμια κατάσταση με δεδομένη την κλιμάκωση των Πούτιν και Ασάντ βλέπουμε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει γρήγορα. Και τελευταία πρόταση κύριε Πρόεδρε. Μόνο από κοινού ως Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι από αυτή την καταστροφική κατάσταση. Μόνο με αλληλεγγύη θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και πραγματικά η δικιά σας η ομιλία ήταν βάλσαμο από την πλευρά του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το EFTD η κυρία Winberg. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στέφαν Λεβέν, είπατε ότι η Σουηδία με αφέλεια υποδέχτηκε τους πρόσφυγες. Προφανώς ε, είσαστε κληρονόμοι της προηγούμενης κυβέρνησης της ε, μετα... μεταναστευτικής πολιτικής. Αλλά εδώ και 1,5 χρόνο εσείς είσαστε υπεύθυνο και τα όσα κάνατε επιβάρυναν την κατάσταση. Η μεταναστευτική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής κυβέρνησης όμως ε, δημιούργησαν χάος στην οικονομία και στην πολιτική. Σήμερα θέλετε να επιβάλλετε σε όλη την Ευρώπη τις συνέπειες της δικής σας αφελούς πολιτικής. Ζητάτε από τα άλλα κράτη-μέλη να σας σώσουν, ενώ σήμερα εσείς έχετε ανάγκη και που όλα τέλος πάντων ε, τα κάνατε λάθος. Λέτε στους άλλους να αναλάβουν τις ευθύνε τους και να υπάρξει αλληλεγγύη. Η δική σας κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Και θα πρέπει κανονικά, θα πρέπει κανονικά να σταματήσει αυτό το, αυτή η ροή των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή η κατανομή των, ε, των ε, μεταναστών ε, που είχαμε επιλέξει μπορεί να λειτουργήσει ποτέ. Είναι δυνατόν να αφομοιώσουμε μια τέτοια γιγαντία μάζα μεταναστών. <coughs> Όλο και περισσότερες χώρες απομακρύνονται από το μηχανισμό κατανομής που εσείς ε, θέλατε, εσείς διαφημίσατε κτλ. Στέφαν, σα παρακαλώ, αναλάβετε τι ευθύνε σα παρότι δεν είναι ευχάριστο. Καταλάβετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εδώ μιλήσετε για απέλαση διαφόρων μεταναστών. Πώς ε, θα τα καταφέρετε όταν δεν μπορείτε να διώξετε καν 30 μετανάστες ε, μέσα σε ένα λεωφορείο. Für για την ομάδα της, των Εθνών και της Ελευθερίας, ο κύριος Στούγκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Είχα επισκεφθεί στην στις αρχές του δεκαετία του 1980 την Σουηδία, που ήταν τότε μια υπέροχη χώρα, όμορφη, ασφαλής, με ευημερία. Και Βλέπαμε πως η Σουηδία προχωρούσε πάντα προς τα εμπρός, ειδικά στον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και οι μαθητές είχαν ένα από τα καλύτερα σχολεία στην Ευρώπη και η χώρα ήταν ανοιχτή και με διαφάνεια. Πέρσι ξαναπήγα με τα παιδιά μου στην Σουηδία και σοκαρίστηκα. Τρόμαξα. Πόσο μπορεί να αλλάξει έτσι μια χώρα. Η, χώρη μου, η κόρη μου είναι 12 ετών και έκανε μια εργασία για τη Σουηδία και πρέπει να, τις να πει στους συμμαθητές της πως η Σουηδία είναι η δεύτερη στον κόσμο χώρα στους βιασμούς. Μόνο στο Λεσότο κινδυνεύουν περισσότερο οι γυναίκες. Πάνω από το Μεξικό, την Ιγυρία, τη Ρωσία. Επίσης πρέπει να τους πει ότι η Σουηδική κυβέρνηση παρακρατά και κρύβει πληροφορίες και για να μην τις εκμεταλλευτούν οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Κύριε Πρόεδρε, τρόμαξα πώς είναι δυνατόν μια χώρα να αλλάξει τόσο πολύ με, μέσα σε 30 χρόνια. Με έναν τρόπο μόνο, με την καταστροφική επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και παίρνει μαζί της και την Σουηδία φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίνε οι πολιτικές ελίτ. Τα ξεμεκέ. Ο κ. Μπαλτσό από τις μία γεγραμμένους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέφεν, είχαν, είχε πει ένας εξέχων Σουηδός οικονομολόγος ότι αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη οι Σουηδοί πιστεύουν όλο και περισσότερο σε συντηρητικές αξίες. Εσείς πιστεύετε σε φιλελεύθερες αξίες, αλλά με τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες ετούμενους ασύλου οι οποίοι οδήγησαν τους Δήμους μας και τις κοινότητές μας σε μεγάλες δυσκολίες. Είναι η δική σας απόφαση, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι σε πολλές πόλεις της, της ε, Σουηδίας έχουμε φτάσει πια στο απροχώρητο, δεν δεχόμαστε να έχουμε άλλους μετανάστες. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ε, κουλτούρα μας, δεν θέλουμε να έχουμε παράλληλες κοινωνίες στη χώρα μας. Μιλάτε για δημοκρατία, αλλά δε, ας δεχτείτε το γεγονός ότι οι πολιτικές αποφάσεις γίνονται με τη θέληση του λαού. Στην Ουγγαρία έγινε δημοψήφισμα. Ήταν αυτή μια πραγματικά κυριαρχή χώρα, όχι σαν για εμά. Για το ΕΛΚ, <clears throat> ο κύριος Γκονσάλε Πόνς έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητή. Κύριε Γκονσάλε Πόνς, το μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη που δεν την έχουμε γνωρίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με απάνθρωπου τρόπου δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Με το να κλείσουμε τα σύνορα, να υψώσουμε τύχη, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της, ε, των προσφύγων. Αυτό απλώ κάνει πιο μεγάλη την απόγνωση και πιο μεγάλη την απανθρωπ, απανθρώπιση των Ευρωπαίων. Έχουμε μια μεγάλη δυσκολία ενώπιόν μας και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουμε τον χώρο του Σέγγεν. Οι εθνικές λύσεις δεν μπορούν να λύσουν τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Αντίθετα, <clears throat> οξύνουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρώπη, γιατί σήμερα οι εθνικές λύσεις δεν είναι επαρκείς για να λύσουν ούτε καν τα εθνικά προβλήματα η κυβέρνησή σας αποφάσισε να εφαρμόσει συνοριακούς ελέγχους μονομερός και υποχρεώνει και τις ιδιωτικές μεταφορικές εταιρείες να κάνουν έλεγχο σε αυτούς που μεταφέρουν. Παραγματικά χάρη η κυβέρνησή σας είπε ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την ε, αναστολή του Σέγγεν για τρία χρόνια, όταν οι κανόνε επιτρέπουν μόνο για δύο χρόνια μια τέτοια αναστολή. Αυτέ είναι εθνικέ αμυντικέ λύσει, οι οποίε είναι σαφώ ανεπαρκεί. Μπορεί να είναι καλές, ίσως όπως πιστεύετε εσείς για τη Σουηδία, είναι σίγουρα κακές για την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν πάρα πολλοί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντίον της ε, συμφωνίας με την ε, Τουρκία. Εσείς όμως Θέλετε αυτή τη στιγμή να υψώσετε τύχη και να κρατήσετε έξω του πρόσφυγε. Λοιπόν, ποιο είναι πραγματικά πράσινο, ποιο είναι πραγματικά ευρωπαϊστή. Όταν σταματάμε να οικοδομούμε την Ευρώπη, ανασωπηρώνεται ο εθνικισμό και με τον αθνικισμό πάντα και η ξενοφοβία. Πάντα ο εθνικισμό οδηγεί σε λαϊκισμό και φανατισμό. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη στην πολυμορφία, όπως είναι και το σύνθημά μας. Σήμερα πρέπει να είμαστε πραγματικά ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ζητήσατε μια πιο κοινωνική Ευρώπη, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σα όσο θέλετε μια Ευρώπη η οποία να είναι κοινωνική, όταν αντιμετωπίσετε ένα πραγματικό ε, πρόβλημα κοινωνικό όπως είναι αυτό των μεταναστών, δεν μπορείτε να ορθώνετε τύχη και να κλείνετε τα σύνορά σα. Αυτό μόνο οι λαϊκιστές θα το κάνουν. Για την σοσιαλδημοκρατική ομάδα η κυρία Ούλσκοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Λέβεν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Είναι πολύ θετική η παρουσία σας. Ακούσαμε τις παρατηρήσεις σας. Ακούσαμε και κάποιες αδικαιολόγητες ε, δηλώσεις από ορισμένου συναδέλφους. Πολύ συχνά μου συμβαίνει αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό που βρίσκεστε εδώ πέρα. Όσον αφορά το ζήτημα τη ανισότητα, μια ανισότητα η οποία αυξάνεται όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 23 εκατομμύρια είναι τα άνεργα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια αυτή είναι τα, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Και ορισμένοι ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λέγανε ότι υπό αυτών των συνθήκων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή της ανεργίας, θα έπρεπε να έχουμε χαμηλότερους μισθούς και λιγότερο προσταυτικές εργασιακές συνθήκες. Πολλοί ουσιαστικά ζητούν μια κατακαιρματισμένη αγορά εργασία και πολλέ φορέ κατακαιρματισμό ανάμεσα στου Ευρωπαίου πολίτε που εργάζονται και του νεοαφιχθέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα εργάζονταν σε χειρότερε εργασιακέ συνθήκε. Με αυτό, όπω καταλαβαίνετε, θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανισότητα. Εμεί είμαστε σοσιαλδημοκράτε. Δεν θέλουμε άλλο κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν θέλουμε άλλο ντάμπινγκ όσον αφορά του μισθού. Δεν θέλουμε ανταγωνισμό ο οποίο να βασίζεται σε χαμηλότερου μισθού και σε όλο και επιδεινόμενε εργασιακέ συνθήκε συνθήκε. Καταλαβαίνετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε σε μία δίνη που φέρνει σε όλο και δυσκολότερη θέση του Ευρωπαίου πολίτε. Δεν θέλουμε εργασιακό και κοινωνικό ντάμπινγκ, θέλουμε ισότιμη αμοιβή για ισότιμε θέσει εργασία, αλλά πραγματικά μπορούμε να βασιστούμε στη δήλωση αυτή που έκανε ο κύριο Γιούγκερ. Είμαι σίγουρο ότι πιστεύει αυτά τα οποία λέει, αλλά μπορεί πραγματικά να κάνει τα λόγια του πράξη. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτική και γι' αυτό το λόγο καταφεύγουν σε ακροδεξιά κόμματα μοιάζει με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, σαν αυτούς που έχουμε στην ε, χώρα μας. Και πολλές φορές τα πράγματα είναι και ακόμα χειρότερα. Πάρα πολλοί λοιπόν στρέφονται προς ακραία κόμματα πρόκειται για ψηφοφόρου που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαντά πλέον στα πραγματικά του προβλήματα με ουσιαστικέ λύσει. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε τα προβλήματα αυτά, θέλουμε να δώσουμε τέλο στο κοινωνικό dumping, πρέπει να το κάνουμε το στομότερο δυνατό. Διαφορετικά όσο καθυστερούμε θα σπρώχνουμε όλο και περισσότερου πολίτε προ ακραίε θέσεις. Ακούσαμε χθε διάφορα μέτρα όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη. Είπαμε ότι ε, Όλο και περισσότερο κοινωνικοί εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερες αρμοδιότητες Πιστεύετε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα καταφέρουμε να έχουμε πραγματικά ισότιμες αμοιβέ για τις ίδιε θέσεις απασχόλησης Για τους φιλελεύθερους έχει το λόγο ο κ. Φέντερλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πρωθυπουργέ Στέφαν Λεύθεν. Ήρθατε σε αυτό το κοινοβούλιο σε μια κάπως δύσκολη χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την πρόκληση κλιματικής αλλαγής, την ανάγκη να βρούμε λύσεις για το μέλλον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως και το προσφυγικό πρόβλημα, να βρούμε τις λύσεις σε όλα αυτά. Και επιπλέον έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι απασχολησμένη με τη συζήτηση για το Brexit και όλο και περισσότερο κλειδονίζεται από το λαϊκισμό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Πρωθυπουργέ, με το να σας επενέσω Σπάνια ήσασταν τόσο σαφείς όπως σήμερα για αυτά που είπατε. Είπατε για κοινέ αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν συμπεράσματα και συνέπειες. Πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος παίζει ηγετικό ρόλο για τα θέματα αυτά. Χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Αλλά συγχρόνως βλέπουμε τι γίνεται στο Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις και μετά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα γίνει ένα αδύναμο, ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτη ανικανότητα. Ποιο είναι το νόημα του να έχουμε ένα συμβούλιο, αν η αποφάση του δεν συμβούλιο μεταναστεύσεων, ήταν μία από τις περιπτώσεις όπου πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι λιμένες αποφάσεις εφαρμόζονται. Έχω και κάποιες αφιβολίες για την έννοια της κοινωνικής Ευρώπης που αναφέρετε κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς δεν συζητούσατε με τον Ντέβιτ Κάμερον και στις συνομιλίε αυτές ουσιαστικά θάψατε κάτω από τη γη την κοινωνική Ευρώπη. Δεν κάνατε κάποιες υποσχέσεις στην προεκλογική εκστρατεία εναντίον αυτής της έννοιας. Μάλλον υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης, αλλά πώς συνδέεται αυτό με τις δηλώσεις που κάνατε μαζί με τον ε, David Cameron. Έχει χάσει το δρόμο της η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Τι είναι να συμφωνώ με τον κύριο Χέρκμαρκ ότι οι σοσιαλδημοκράτες που έφεραν την Σουηδία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πάρσον, ο οποίος ζήτησε την ε, διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον κύριο Σβάινφελτ, ο οποίος ενίσχυσε τη συνεργασία, ήταν πάντα ευρωπαϊστές. Εσείς όμως τι πιστεύετε για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Για την ομάδα της ΓΚΟΕ το λόγο έχει η πρόεδρος Τσίμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν θεωρούσα ότι θα ήταν δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχουν τέτοιε εκπλήξει. Ένα βουλευτή από την άλλη, από του φιλελεύθερου, να θέσει ακριβώ τα ερωτήματα που εγώ ήμουν έτοιμη να σα θέσω. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε από κοινού να αντεπεξέλθουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μονάχα άμα έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μα. Αυτό σημαίνει όμω επίση ότι ναι, χρειαζόμαστε την κοινωνική Ευρώπη. Εσείς όμως είστε και μέλος του Συμβουλίου και συνυπεύθυνος για την συμφωνία η οποία έγινε με την Μεγάλη Βρετανία που ουσιαστικά θέτει σε δοκιμασία την κοινωνική Ευρώπη και ουσιαστικά είναι μια υπαναχώρηση σε σχέση με την έννοια της ευρωκοινωνικής Ευρώπης. Το να ανατραπούν σημαντικοί κανονισμοί που είχαμε σε σχέση με την ε, ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη κρίση για την Ευρώπη. Μερικοί από αυτούς τους τόσο σημαντικούς πυλώνες των βασικών ελευθεριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα ακυρωθούν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μου φαίνεται πολύ ανησυχητικό. Επίσης, όταν λένε οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μια αντίφαση, από τη μια μεριά λέτε θέλουμε κοινωνική Ευρώπη, από την άλλη πλευρά λέτε ότι θέλετε μια κοινή λύση για το θέμα των προσφύγων, αλλά στην πράξη δεν το κάνετε αυτό, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν δεν μπορούμε να έχουμε κοινή αντιμετώπιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τους πρόσφυγες επί τη βάση της προέλευσής τους, της χώρας, της πόλης από την οποία έρχονται. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την συναδελφό μου τη Μαριον Μπιόρκ. Περιμένουμε από εσά εσείς συγκεκριμένα να κάνετε την απαραίτητη αυτή κίνηση όπως ζητήσατε και στις συζητήσεις για τον αφοπλισμό. Μπορεί να θέλουν όλοι να κάνουν κάτι, αλλά κάποιο πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Κάντε και εσεί τα απαραίτητα για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για τα θέματα αυτά. Για την πράσινη ομάδα, ο κύριο Έριξον έχει το λόγο. Η κυρία Έριξον. Κύριος. Κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, βεβαίω η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ε, Τουρκίας ε, αφήνει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Βεβαίως είναι καλό πράγμα ε, που η Σουηδία μίλησε για την τήρηση των διεθνών κανόνων για το άσυλο. Πώς αυτά βεβαίως θα εφαρμοστούν δεν είναι σαφές και έχω μερικέ ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω στον Πρωθυπουργό. Νομίζετε ότι η Τουρκία θεωρείται ασφαλή χώρα η Σουηδία δεν το πιστεύει αυτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή θέση σε σχέση με το θέμα αυτό. Είδα αλλιώ ε, θα είναι ε, κάτι άλλο που θα προσδιορίσει αν θα επιστραφούν οι μετανάστες και όχι από που προέρχονται ή αν έχουν καλή αίτηση ασύλου. Αν η οδός η ελληνική κλείσει, τι άλλες οδούς θα διαλέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ασφαλέστερες ε, και είσαστε βέβαιος ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι μια συμφωνία συμφωνία που θα επιδεινώσει την κατάσταση. Επίσης, τι γίνεται με την Σουηδική κυβέρνηση πώς στο μέλλον θα ε, αντιδράσετε σχετικά με αυτά τα ζητήματα για να μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αρχίζει να εφαρμόζει το δικαίωμα ασύλου. Ξέρετε πώς θα εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό στο μέλλον. Και μια προσωπική ερώτηση. Εσείς προσωπικά μετά από όλες αυτές τις συμφωνίες, όλες αυτές ε, τις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις έχετε καμιά ελπίδα απέναντι στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζετε ότι θα τις υποχρεώσεις και θα γίνει μια δίκαιη κατανομή ε, των μετανοστών βασιζόμενη στην αλληλεγγύη. Τώρα για την ομάδα FNDD, ε, κύριος Λούντγκρεν. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, να είμαστε λοιπόν επιτέλους ε, εδώ κανονικοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, απλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά πιστέψαμε κάποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστέψαμε στο ειδικό μοντέλο, ανήκαμε στην δικαλιστική οργάνωση μεταλλορίχων, αλλά εδώ πέρα τελειώνει τελικά η ρόδινη αυτή ιστορία. Θεωρώ ότι ήσασταν πάρα πολύ αφελεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Κάνετε πάρα πολλά λάθη και εγώ και εκπρόσωποι του δικού μου κόμματο για πάρα πολύ καιρό είχαμε πει ξεκάθαρα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, ποια θα ήταν η έκβαση αυτή τη πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενε κυβερνήσει τη Σουηδία. Η αφέλεια αυτή θα οδηγούσε σε τραγικά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια γελία κατάσταση, το θέτω έτσι, και ορισμένε από τι δηλώσει που κάνατε σήμερα ουσιαστικά αντιστοιχούν ακριβώ αυτό. Πραγματικά ήσασταν πάρα πολύ υποκριτή. Διατηρήσατε μια ιδιαίτερη υποκριτική στάση. Η Γερμανία σαφώ ευθύνεται για την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε όμως τι γίνεται και στι διάφορε νομαρχίες τη χώρα μου. Ένα 60% των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι οικονομικοί μετανάστες και από την άλλη έχουμε 16.000 παιδιά τα οποία χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στον κόσμο ακριβώς επειδή δεν έχουν ε, φρέσκο νερό, πρόσβαση σε τρόφιμα. Θεωρώ ότι είναι τρελή κατάσταση αυτή. Στέφαν είπατε ότι είστε ικανοποιημένος με τη συμφωνία που συνάφθη με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς, η κυβέρνησή σας θα ζητήσετε κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο ζήτησε και πήρε τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει πάρα πολλά χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα ζητούσετε και εσείς κάτι το ανάλογο. Πραγματικά κατηγορώ την πολιτική ορθότητα της κυβέρνησης αυτής. Σας ευχαριστώ. E Ο κύριος Μάιερ για την ομάδα ENF. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Δεν θα μείνει πέτρα λίθος επιλίθου στην Ευρώπη. Έχουμε διαβάσει όλοι τα σχόλια και εγώ είδα κάτι που μου το έδωσαν οι φοιτητέ μου. Όταν ακούω τη συζήτηση και αυτά που λένε οι συνάδελφοι, η κυρία Χάρμς, η κυρία Βιόρκ, ακόμα περισσότερο με εντυπωσιάζει. Αυτές οι κυρίες λέω ζουν σε άλλο πλανήτη από τους υπόλοιπους εμάς. Όλα αυτά τα οποία ακούμε εδώ πέρα είναι μια επικίνδυνη αφέλεια. Αν δούμε λοιπόν αυτή την κρίση μετανάστευση η οποία είναι εξελίξη και η οποία αντιμετωπίζεται με ανεγκέφαλο τρόπο και με τελείως με τέλεια έλλειψη οργάνωσης και ήρμου βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοιο πολιτικό λόγο έχουν βοηθήσει να ενισχυθεί αυτή η κρίση και να οξυνθεί περισσότερο. Ενώ συγχρόνως η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι τα μεμονωμένα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν σωστά τις αρμοδιότητές τους είναι πολύ πιο ικανά να λύσουν τα προβλήματα από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε αυτό ήδη στην Αυστρία, ότι η κυβέρνηση δέχεται ιδέες όπως η ιδέα του ένα προς ένα. Ακολουθεί τέτοιες ιδέες. Η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, Μέρκελ μας έχει ρίξει σε μια βαθιά κρίση και η μόνη λύση, η μόνη δυνατότητα λύση που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά από τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μεμονωμένες. Έχουμε πολλά αδικήματα που έχουν γίνει από μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική στην Αυστρία. Το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι 75% αυτών οι οποίοι ζητούν άσυλο είναι άνδρες και αυτά μας θυμίζουν γεγονότα που είναι αρνητικά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο, να μην μπορούν οι γυναίκες να κυκλοφορούν ανενόχλητες στο δρόμο. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Βίκτορ Όρμπαν γιατί τουλάχιστον έχει κερδίσει τον πρώτο γύρο και έχει εμποδίσει αυτή την απόλυτα λανθασμένη συμφωνία με την Τουρκία. Ο κύριος Φουντούλης από τις μία γεγραμμένους. Δυστυχώ η σημερινή κατάσταση στην ευρωπαϊκή ένωση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η καλύτερη. τα προβλήματα είναι πολλά και αντί να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσει με συνεχείς αναβολέ και καθυστερήσει, συσσωρεύονται ακόμα περισσότερα. ειδικότερα στι χώρε του νότου η ανεργία η ανεργία των νέων οι περικοπέ μισθών και συντάξεων η κατάρρευση του συστήματο υγεία είναι πολύ σημαντικά θέματα. στην ατζέντα των θεμάτων προεξέχουν το μεταναστευτικό και το οικονομικό και έχουμε εστιάσει εκεί αγνοώντας άλλα εξίσου σημαντικά για τα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις. ιδεολογικές αγκυλώσεις και σκοπιμότητες πολιτικών ομάδων που είχαν μάθει να μην ακούγονται διαφορετικές φωνές και απόψεις υπονομεύουν τόσο το αίσθημα δημοκρατίας όσο και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού άλλων πολιτικών απόψεων. στη δημοκρατία δεν υπάρχουν μέτρα και κόκκινες γραμμές. δεν ζυγίζουμε περισσότερη ή λιγότερη δημοκρατία. οι ιδεολογίε στην ευρώπη υποτίθεται ότι δεν διώκονται όπως και οι διαφορετικές απόψεις η ιστορία για κάποιες χώρες έχει γραφτεί και δεν εξοραίζεται όπως επιθυμούν κάποιοι. γι' αυτό θα πρέπει να μην ξεχνάμε το παρελθόν για να βαδίσουμε στο μέλλον. σαν ευρωπαϊκή ένωση ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρντίνη απο το θα ήθελα να συζητήσω ζητήσω κάποιες εξηγήσει, γιατί εσείς είστε υπέρ του PNR στο Συμβούλιο, έτσι δεν είναι. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δύο στο Κοινοβούλιο που το απορρίπτουν. Αναφέρομαι στον κατάλογο ονομάτων των επιβατών. Επίσης, πώς μπορούμε να περάσουμε ποτέ από μια πολιτική ανοιχτών θυρών σε μια πολιτική κλειστών θυρών που ουσιαστικά αντιβαίνει στις βασικές αρχές των σοσιαλδημοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι ακόμα κύριε Πρωθυπουργέ, πώς είναι ποτέ δυνατόν ακόμα και στην Σουηδία που είναι χώρα πρότυπο υποδοχής και ισότιμων ευκαιριών αυτή τη στιγμή να έχουμε το δραματικό φαινόμενο του αντισημιτισμού. Ακόμα και στο Μάλμο, μία πόλη η οποία δέχτηκε χιλιάδες Εβραίου στο παρελθόν προσπαθούσαν το 1943 να γλιτώσουν από τον ναζισμό, είδαμε πάρα πολλά φαινόμενα και πάρα πολλά κρούσματα μη ανοχή. Και υπάρχουν ακόμα πολλέ εκατοντά, εκατοντάδε Εβραίοι που ζουν εκεί, σύμφωνα με μια εκπομπή που είδα στην τηλεόραση, και μάλιστα φοβούνται πάρα πολύ να βγουν ακόμα και από το σπίτι του. Βέβαια, στο κόλμη τα πράγματα μπορεί να είναι εντελώ διαφορετικά, πάντω όλα αυτά μα προκαλούν ανησυχίε. Πέρα από τα πολλά, πολύ ωραία λόγια που μα είπατε σήμερα, πείτε μου πραγματικά τι προκύπτει να κάνει η δική σα η κυβέρνηση γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Αν πραγματικά, κύριε Πρωθυπουργέ, οι Εβραίοι που έχουν συμβάλει τόσο πολύ στον ευρωπαϊκό πολιτισμό αρχίζουν πλέον να θεωρούν ότι ακόμα και η Σουηδία δεν είναι σπίτι τους, είναι μια χώρα στην οποία φοβούνται να ζούνε, τότε πραγματικά δεν υπάρχουν πλέον πάρα πολλές ευίωνες ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Ροντρίγιος, για τους σοσιαλδημοκράτες έχει το λόγο. Μεγάλη τιμή κύριε ε, Πρωθυπουργέ και χαρά να σας υποδεχτούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλάτε με μια στεντόρια ευρωπαϊκή φωνή βασισμένη στη σουηδική εμπειρία. Η Σουηδία έχει βέβαια προβλήματα, αλλά είναι ένα από τα φωτεινά παραδείγματα τα οποία μπορούν να ακολουθηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία, όπως ήδη αναφέρθηκε έχετε πολύ υψηλά πρότυπα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Σουηδία. Δεύτερον, η Σουηδία είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να αγωνιστούμε για βιώσιμη ανάπτυξη με μια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική διάσταση συνάμα και περνάτε τώρα μια φάση ισχυρής ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Επίσης, η Σουηδία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα διεθνούς υπευθυνότητας. Και επίσης, παρά τα προβλήματα που έχει η Σουηδία, η Σουηδία παραμένει ένας πολύ σημαντικός εταίρος, ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα του πώς να ενσωματωθούν στην κοινωνία σας οι πρόσφυγες. Εγώ πήγα πάλι στη Σουηδία και αυτό το οποίο είδα πρέπει να πληροφορήσω την Ολομέλεια για αυτό. Η Σουηδία εξακολουθεί να διαχειρίζεται μια πολύ μεγάλη ροή προσφύγων. Και είδα για πρώτη φορά να είναι μια αξιοπρεπής υποδοχή στα σύνορα των προσφύγων. Είδα μετά την κατανομή των προσφύγων σε όλη τη χώρα. Σε πολλούς δήμους και πόλεις όπου μπορούσαν να βρουν στέγαση και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Και επίσης να συμμετάσχουν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης για να ενσωματωθούν στην τοπική οικονομία. Αυτή ήταν η πραγματικότητα λοιπόν που εγώ είδα στη Σουηδία. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτά είναι πολύ απλά αλλά πολύ ανθρώπινα μέτρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ρεύματος και τα οποία θα πρέπει να γίνουν σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ και πάλι. Τελευταίος ομιλητής έχει το λόγο ο κύριος Άντερσον από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται εδώ. Ελπίζω ότι βρήκατε την συζήτηση αυτή ενδιαφέρουσα και παραγωγική. Μιλάμε για μια κοινωνική Ευρώπη, αλλά δεν αναφέρατε το στοιχείο αυτό, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ευρωζώνη που δεν λειτουργεί καλά και που συνέβαλε σε αυτήν την οικονομική κρίση και στην μεγάλη απασχόληση. Είναι προφανές ότι η Σουηδία ε, πήρε την σωστή απόφαση όταν δεν θελήσαμε να προσχωρήσουμε στην ΟΝΕ με δημοψήφισμα. Ακούω όμως πολλούς συναδέλφους εδώ ε, να λένε ότι η Σουηδία δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίζει επαόριστον έτσι να απέχει από την ΟΝΕ διότι αλλά εμείς τηρούμε την επιλογή του λαού. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα ίσως σκεφτούν ότι θα ήταν καλό για την Σουηδία να έχει μια εξαίρεση που να αναφέρεται στις συνθήκες, ένα opt-out. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες σε όλες τις χώρες που δεν θέλουν να προσχωρήσουν στην ΟΝΕ, να υπάρξουν εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις για τις χώρες αυτές. Αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι καλές για όλους, όχι μόνο για τους λίγους. Ελπίζω ότι η Σουηδία θα τεθεί επικεφαλής αυτής της προσπάθειας για να υπάρξουν αυτές οι συνθήκες. Ο Πρωθυπουργό τη ε, Σουηδίας, ο κ. Λεύτουεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση και για όλες τις παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω την άποψή μου για τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, στον Γκαρανθερ Μάικ, εγώ ε, δεν θέλω να υπάρξουν πάρα πολλά νέα μέτρα που θα επιβαρύνουν τις εταιρείε. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι έχουμε μια κοινή οικονομία. Έχουμε μια κοινή αγορά εργασίας και σε αυτή την αγορά εργασίας χρειαζόμαστε ένα μέλλον για αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που παράγουν, παράγουν το πλούτο ε, που εμείς κατανέμουμε. Και δεν ε, βλέπω πώς μπορούμε ε, να πούμε ότι θα είναι αρνητικό το μέλλον, ότι θα μειωθούν οι μισθοί, ότι οι όροι εργασίας θα επιδεινωθούν. Αυτό δεν είναι το μέλλον που οι ευρωπαϊκοί λαοί προσδοκούν. Έχουμε με μια κοινό συμφέρον, μια κοινή ευθύνη να ε, εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας θα διέπεται από κοινέ αξίες και βεβαίως οι διάφορες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, κυβερνούν με τον τρόπο που πιστεύουν κατάλληλο. Είδαμε το 2007 ε, την περίπτωση Λαφάζ, είδαμε ότι ότι τα συνδικάτα της Σουηδίας δεν μπορούσαν να εξαρτηθούν από τις συλλογικέ συμβάσεις. Αυτό ήταν εσφάλμα, θα ήταν εύκολο να πούμε ότι αν υπάρχουν ε, ε, συλλογικές ε, συμβάσεις θα πρέπει να τηρηθούν εφόσον δεν υπάρχει διάκριση. Αλλά οι εργαζόμενοι της Ευρώπης παρακολουθούν την κατάσταση και βλέπουν ότι το μέλλον θα είναι με χαμηλότερους μισθούς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υπέρ αυτής της συνεργασίας. Ας υποσχεθούμε στους εαυτούς μας ότι θα αναπτύξουμε μια αγορά εργασίας στην Ευρώπη που θα υπόσχεται κάτι καλό για το μέλλον και ας κατανοήσουμε ότι αυτοί οι γυναίκες και άνδρες που πάνε να εργαστούν κάθε μέρα είναι οι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Είναι αυτοί, αυτές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καλές συνθήκες εργασίας και ένα καλό μέλλον. Υπήρξαν επίσης πολλές παρεμβάσεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση, την κρίση των προσφύγων. Το μήνυμά μου είναι το εξής. Έχουμε και θα έχουμε πρόσφυγες στον κόσμο, δυστυχώς. Και το πρόβλημα όπως λένε μερικοί, λένε ότι είναι σουηδικό πρόβλημα. Εμείς δεν προκαλέσαμε το πρόβλημα διότι υποδεχόμαστε πρόσφυγες. Το πρόβλημα είναι στη Συρία. Το πρόβλημα είναι στην Μέση Ανατολή που αναγκάζει τους ανθρώπους να φεύγουν διότι φοβούνται φοβούνται, είναι τρομοκρατημένοι, είναι στο μέσο του πολέμου. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και νομίζω ως ανθρώπινων ότι θα πρέπει να πούμε σε αυτούς που φεύγουν ε, γιατί φοβούνται για τη ζωή τους, ναι πρέπει να σας βοηθήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα που είναι η αιτία της κατάστασης που τους οδηγεί στην φυγή. Υπάρχουν αυτοί που έρχονται δεν μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα. Μερικά, μέρη πιστεύουν ότι πρέπει να κλείσουμε την πόρτα. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε αυτούς που φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Όλοι μαζί, 28 κράτη-μέλη. Και αν το πράξουμε μαζί, αν το πράταμε μαζί θα το είχαμε επιλύσει το πρόβλημα. Δεν θα ήταν πλέον πρόβλημα. Είμαστε 508 ε, εκατομμύρια κάτοικοι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα μαζί. Και μερικοί λένε βεβαίως δεν θα συμμετάσχουμε. Αν επιλέξουν ένα, τη μη συμμετοχή νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι αν δεν συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα, το σύστημα ασύλου, δεν θα πρέπει ίσως να συμμετέχουν και στο σύστημα Schengen. Δεν μπορούν να επιλέγουν μόνο τα καλά πράγματα, τα εύκολα πράγματα. Και στα δύσκολα ε, να φεύγουν. Θα πρέπει να κάνουν και τα πιο δύσκολα, τα πιο λεπτά πράγματα. Εμείς θέλουμε ένα μελλοντικό σύστημα που στην πραγματικότητα να μπορεί να κατανείμει τις ευθύνες μεταξύ των 28. Δεν ξέρω. Μερικοί ε, αντιστέκονται Υπάρχουν αντιδράσεις. Τις ακούω, αλλά αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει καλά, βοηθώντας οι μεν τους δε. Και αυτοί που δεν θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να εξετάσουν και κάτι άλλο. Αν αυτό δεν λειτουργήσει θα επηρεάσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αυτούς οι οποίοι τώρα ε, κάθονται στη γωνιά τους και δεν κάνουν τίποτα. Θα επηρεαστούν και αυτοί. Αν θέλουμε μια, μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική πρέπει να συνεργαστούμε επίσης για αυτά τα δύσκολα θέματα. Αυτό, αυτή είναι η άποψή μου και θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι μεν προς τους δε. Σχετικά με τη συμφωνία με την Τουρκία πιστεύω ότι είναι σωστή, ότι πρέπει να βρούμε μια λύση και να έχουμε συνεργασία με την Τουρκία. Ή αλλιώ ε, δεν θα προχωρήσει το πράγμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις λεπτομερείς ερωτήσεις. Ο πρόεδρος Τούσκ έλαβε μια εντολή να διαπραγματευτεί βάσει των αρχών αυτών θέλουμε αυτή η λαθρέα διακίνηση των ανθρώπων να σταματήσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Διότι όσοι είναι εναντίον όλων των λύσεων πρέπει να μας δείξουν τις αναλλακτικέ λύσεις. Τώρα χιλιάδες άτομα διακινδυνεύουν τη ζωή τους ε, στη θάλασσα. Και έχουμε άτομα τα οποία πουλούν αυτά τα ταξίδια και δεν νοιάζονται, δεν νοιάζονται καθόλου για τη ζωή των ανθρώπων που μεταφέρουν. Έχουμε πάνω από 400-500 άτομα σήμερα που πέθαναν. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό, να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι η μόνη λύση, βεβαίως δεν είναι η μόνη λύση, αλλά είναι μια, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις και με, θα, τότε θα συζητήσουμε το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Επίσης μου τέθηκε ερώτηση για... Ε, για την οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων αν κατάλαβα ε, την ερώτηση αν η οδηγία θα λύσει τα προβλήματα. Όχι, δεν θα τα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα δείξει στους εργαζόμενους και στους εργοδότες της Ευρώπης ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που θα λειτουργεί καλά και που θα τηρεί ε, τις συλλογικές συμφωνίες και τις ρυθμίσεις στις χώρες μας. Ανεξάρτητα από το δρόμο που θα επιλέξουμε ως χώρες θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την πλατφόρμα, αυτή τη δυνατότητα. Για την χώρα μου σημαίνει σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων. Είναι καλός δρόμος, ένας αποτελεσματικός ε, ε, δρόμος με οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή μεταξύ των πολιτών και κατοίκων της χώρας μου. Νομίζω ότι αυτό που πρότεινε η Κομισιό δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ένα βήμα προς τα μπρος και που θα δώσει περισσότερη ελπίδα στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους της Ευρώπης. Και αυτό είναι μια, ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ.